και τις καλύτερες πρακτικές των κρατικών προμηθειών, μειώνοντας τον αντίκτυπο της αγορά. Από κοινού, τα μέτρα αυτά θα παράσχουν σαφή μηνύματα προς την αγορά, επιτρέποντας τις αρχές, τους κατασκευαστές και τους επενδυτές να προγραμματίσουν καλύτερα την μετάβασή μας μέχρι τα μέσα του αιώνα στην κινητικότητα μηδενικής ε, εκπομπής βελτιώνοντας την μείωση της συμμετοχής του άνθρακα στην κινητικότητά μας και την επίτευξη του μηδενικού στόχου το 2050. E Ευχαριστώ, Επίτροπε. Για την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, Ντέλη. Έχει το λόγο που δεν είναι εδώ όμως. Αργότερα. Πολιτικές ομάδες. Ξεκινούμε από το ΕΛΚ. Ο κύριος Πίπερ έχει το λόγο. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η προστασία του περιβάλλοντος και η μείωση των επιζήμιων ουσιών αριθμίζεται καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το εθνικό επίπεδο σε ό,τι αφορά την ε, αποδοτικότητα την ενεργειακή τη μείωση των εκπομπών και έτσι λοιπόν εργαζόμαστε καλύτερα στον οικολογικό σχεδιασμό, στη ενεργειακή επισήμανση και σε πολλά άλλα θέματα συνεργαζόμαστε ευρωπαϊκά. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει τέτοια εγγύηση. Είμαστε υπέρ των ευρωπαϊκών διατάξεων. Δεν θα πρέπει όμως να επισέλθουμε σε μεγάλο επίπεδο λεπτομερίας και κυρίως όχι στους δήμους και στις κοινότητες να μπούμε να κάνουμε κομμάτι με τις διατάξεις αυτές, ε, κυρίες και κύριε, θεωρώ ότι ε, ανοίγουμε ένα μεγάλο πλήγμα στον κόλπο των ε, Δήμων και Κοινωνιτήτων, γιατί απέχουμε πολύ από τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τις ποσοστώσεις για τα ηλεκτρικά ε, λεωφορεία, κάνουν τις μεταφορές πολύ ακριβές και το πώ ε, ρυθμίζονται όλα αυτά. Θα πρέπει να τα αφήνουμε στο ε, επίπεδο των τοπικό. Όχι να υπάρχουν ε, γενικές από τις Βρεξέλλες και στην πατρίδα μου θα υπάρξει μεγάλη αντίδραση και δικαίω για την υπερβολική ανάμειξη των Βρυξελών και μεγάλο τμήμα του ΕΛΚ θα απορρίψει την οδηγία αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Και το λόγο λοιπόν τώρα έχει από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες ο κύριος Ντάνς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Τις ευχαριστίας μου στον εισηγητή, τον κύριο Γκριπ και την Κομισιόν. Το Συμβούλιο Κρίμα δεν είναι εδώ. Εξαιρετική δουλειά που έχουμε κάνει. Κύριε Κρύπ, είσαστε πολύ δίκαιος ως εισηγητής πολύ αμερόληπτος. Ε, διεξάγατε τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των διαφορετικών ομάδων με εξαιρετικό τρόπο. Συγχαρητήρια. Ο φάκελος αυτός είναι πολύ καλό παράδειγμα για το λόγο για τον οποίο έχουμε εκλεγεί εδώ και το ρόλο μας. Πρέπει να γίνουμε πιο δραστήριοι στον καθαρισμό των οχημάτων, στο να κάνουμε τα οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους πιο καθαρά όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και γιατί ε, η ποιότητα γενικότερα του αέρα τη πόλη είναι πολύ κακή. Οι κρατικέ προμήθειε αντιπροσωπεύουν το 14% του ΑΕΠ τη Ευρωπαϊκή και το 45% των ε, λεωφορείων που κυκλοφορούν. Είναι λοιπόν πολύ σωστό και πολύ επίκαιρο που θα χρηματοδοτήσουμε τα πιο φτηνά, ε, πιο συγγνώμη, καθαρά οχήματα ε, μέσω των κρατών μελών. Το 2030 το 60% των λεωφορείων θα πρέπει να πληρούν τους όρους οδηγίας. Η Κομισιόν βέβαια και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι τοπικές αρχές θα έχουν τα κατάλληλα μέσα και επαρκείς πόρους. Απαντώντας στους συναδέλφους του ΕΛΚ θα ήθελα να πω το εξή. Χρειαζόμαστε αυτή τη φιλοδοξία. Δεν μπορούμε να καθόμαστε στον καναπέ μας και να ελπίζουμε ότι τα πράγματα από μόνα τους κάπως θα κινηθούν. Πρέπει να πάρουμε δύσκολε αποφάσεις σήμερα σε όλα τα κράτη-μέλη βλέπουμε νέου να διαδηλώνουν, να διαμαρτύρονται και όχι μόνο νέου γενικότερα ευαισθητοποιημένου πολίτε. Θα πρέπει να αντιδράσουμε τώρα. Και είμαι περήφανο που το κάνουμε. Το Κοινοβούλιο και οι πόλει είναι αυτέ που ζητούν πάντοτε περισσότερα, ενώ τα, οι κυβερνήσει, οι κεντρικές κυβερνήσεις είναι αυτέ που κρατάνε τα χαλινάρια. Αυτή είναι η εμπειρία μου τα τελευταία πέντε χρόνια. Ε, δεν ξέρω αν θα επιστρέψω στο κοινοβούλιο αυτό ω Βρετανό. Αν όμω αυτή είναι η τελευταία μου ομιλία, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είστε εδώ για να κάνετε το ορθό. Έμαθα πολλά από εσά και ελπίζω θα επιστρέψω για να μάθω περισσότερα. Thank you very much, dear and good luck. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Καλή τύχη σας εύχομαι. Και τώρα το λόγο έχει από το ECR ο κύριος Ντε για 1,5 λεπτό. Μάρκα, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία Επιτροπή, συνάδελφοι, πριν από λίγο συζητήσαμε για τι πρώτε μειώσει των διοξιδίτων ανθρακά για τα βαρέα οχήματα. Και τώρα έχουμε ένα φάκελο για τα καθαρά και ενεργειακώ αποβατικά οχήματα και πώ θα μπορούμε να τα προωθήσουμε. Είναι καλό το αποτέλεσμα και νομίζω πάρα πολύ σημαντικό ως μήνυμα για την τελευταία ε, ολομέλεια αύριο, την ψηφοφορία δηλαδή, τη τρέχουσα θητεία θα έχουμε δύο φορέ την ευκαιρία να επιλέξουμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα για την καταπολέμηση τη αλλαγή του κλίματο. Στην ε, καταπολέμηση τη ρήπανση τη ατμόσφαιρα, οι δημόσιε συμβάσει αποτελούν όντω ένα σημαντικό κίνητρο για την μετάβαση σε μια κινητικότητα χαμηλών εκπομπών. Οι αρχές θα πρέπει να δράσουν ε, υποδειγματικά και η δική μου κυβέρνηση, η φλαμανδική ε, κυβέρνηση είναι υπέρ μια τέτοια βιώσιμη πολιτική. Χρειάζεται λοιπόν η μετάβαση αυτή για την ε, καταπολέμηση τη αλλαγή του κλίματο, αλλά και για την ποιότητα τη ατμόσφαιρα στι πόλει μα και στι κοινότητέ μα και κυρίω στη χώρα μου. Για την, ε, το κόμμα μου, για το NVA, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξουν στην συμφωνία τεχνολογικά ουδέτερες λύσεις, όχι μόνο οχήματα με μπαταρίες και ηλεκτρικά, αλλά υβριδικά με ε, υγροποιημένο αέριο κτλ. Χρειαζόμαστε όλες τις δυνατότητες για να μπορέσουμε να κινηθούμε πραγματικά προς μια κινητικότητα χαμηλών εκπομπών. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ συνάδελφε. Και τώρα από την Άλτε, το λόγο έχει η κυρία Μιλμπάου Μαραντίκα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ, Θέλω να συγχαρώ καταρχήν τον εισηγητή και όλους τους κοιόδης εισηγητές. Αυτή η πρόταση πρέπει να δώσει δύο βασικά χαρακτηριστικά στον κοινό μας στόχο της μείωσης των εκπομπών στις μεταφορές κατά 20% μέχρι το 2025. Ε, δύο βασικά χαρακτηριστικά, ρεαλισμό και σαφήνεια. Και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα για να ε, σχετικοποιήσουμε τα όσα λέγονται για τον δίζελ. Γιατί μας, ε, το δίζελ ε, μας εμποδίζει να μειώσουμε ε, το, τις εκπομπές, περιμένοντας τις μηδενικές εκπομπές και δημιουργεί μεγάλο κοινωνικό κόστος, διότι ήδη βλέπουμε μείωση στις, στην απασχόληση εξαιτία της κρίσης του δίζελ. Και υπάρχουν εναλλακτικέ που είναι πολύ πιο καθαρές από τον δίζελ. θα πρέπει η μετάβαση να γίνει σταδιακά προς τι μηδενικές εκπομπές θα πρέπει να μπορούμε με ρεαλισμό να καθορίσουμε σαφείς στόχους για το μέλλον. Άλλες ε, χώρες, στους οποίους πουλούν οι δικοί μας κατασκευαστές, το έχουν ήδη κάνει. Προβλεψιμότητα και ρεαλισμός ε, θα πρέπει να βοηθήσουν και τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις να ε, διοχετεύσουν τις επενδύσεις τους με τρόπο έτσι ώστε να αποδώσουν στο μέλλον. Γι' αυτό το λόγο αυτό το κείμενο πέραν το ότι θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα της κρίσης της πωλήση, θα βοηθήσει, θα ενθαρρύνει μια βιομηχανική πολιτική προς τα οχήματα μηδενικών εκπομπών. Επίσης, ε, θα επιτρέψει σε κάθε τύπο μεταφοράς να προσφέρει ό,τι μπορεί σε ό,τι αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα, ε, την κοινωνική αποδοτικότητα και την περιβαλλοντική αποδοτικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, η εμφάνιση νέων τύπων πρόσβασης στα οχήματα. Για παράδειγμα, σε ορισμένε ε, χώρες, όπως τη δικιά μου, ο μέσος όρος ηλικία των αυτοκινήτων από 8 έτη το 2007 πέρασε στα 12,4 το 2017. Το 62% μάλιστα έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 10 ετών. Και θα φτάσει και μερικέ φορέ στα βαν, στα μικρά επαγγελματικά οχήματα, φτάνει τα 13 έτη. Το να μπλοκάρουμε την ανανέωση του στόλου περιμένοντα τα οχήματα μηδενικών εκπομπών είναι πολύ κακό, θα ήταν πολύ κακή είδηση και για το περιβάλλον και για την οδική ασφάλεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, για την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά ο κύριος, η κυρία Κονέτσινα, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε, δεν είμαι πολύ ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Ποιο είναι πραγματικά το αποτέλεσμα αυτό. Υπερβολικές απαιτήσει στους παραγωγούς για τη μείωση των εκπομπών και τίποτα άλλο. Το κείμενο της οδηγίας για την πρόθεση των ε, αποδοτικών οχημάτων ε, θα έπρεπε να οδηγεί σε μια αγορά ελεύθερων ε, καθαρών οχημάτων, αλλά έχει φτάσει πάρα πολύ αργά και περιλαμβάνει πολλά παραθυράκια. Οι, οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει να δαπανίσουν εκατομμύρια ευρώ για να αναπτύξουν αυτές τις τεχνολογίες, αλλά ποιος θα τις αγοράσει ο κρατικός τομέας ε, δεν είναι έτοιμος ακόμα. Τα κράτη-μέλη μεταθέτουν το φορτίο και το κόστος στους κατασκευαστές. Στην πραγματικότητα δεν θα επιτευχθεί μείωση εκπομπών. Τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς επίσης δεν ήταν ικανοποιητικά. Η, η περίοδος μεταγραφής είναι πάρα πολύ μικρή, δεν είναι ικανοποιητική το Κοινοβούλιο πούλησε το θέμα αυτό πολύ φτηνά. Δεν μπορώ να στηρίξω αυτό το κείμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον τελευταίο ομιλητή, είναι η τελευταία φορά, θα σας πω, που προεδρεύω στην Ολομέλη αυτή, αυτή τη θητεία. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την δυνατότητα που μου δώσατε εσείς οι πολλοί και οι λίγοι εδώ σήμερα να είμαι αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου. Κατά τη διάρκεια της θητεία μου προσπάθησα να τιμήσω την θέση αυτή με συμμετοχή, δέσμευση και βούληση να υλοποιήσω τις δεσμεύσεις που είχα αναλάβει όταν ε, προσπάθησα να επαναφέρω τον πλουραλισμό μέσα στο Προεδρείο. Ευχαριστώ λοιπόν όλους σας κβάθους καρδίας και ε, καλή επιτυχία σε όλους όσοι κατεβαίνουν στις εκλογές για να βελτιώσουν την Ευρώπη προς όφελος όλων των πολιτών της Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Για τους ε, πράσινους, ο κύριος Μαρτσελέζη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως έλεγε χθε η Γκρέτα Τόμπεργκ, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο το σπίτι μας ε, ε, καταραίει. Αυτό έχουμε μπροστά μας μια κλιματική κρίση και χρειάζεται σήμερα, χτες μια λύση. Ο, ο, ο κλάδος των οδικών μεταφορών είναι από τους πιο ρηπογόνους. συμφωνούμε σήμερα να βελτιώσουμε την κατάσταση ζητώντας από όλα τα κράτη-μέλη ε, να αντιμετωπίσουν χρησιμοποιήσουν το 20% των οχημάτων με, κα, με καθαρότερο τρόπο. Αυτό σίγουρα είναι βελτίωση. Ωστόσο, όπως θύμισε χτες η Γκρέτα Τόμπεργκ, μπροστά στην κρίση δεν προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, αλλά ό,τι είναι δυνατό. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια πραγματική επανάσταση στον κλάδο των μεταφορών και της κινητικότητας, μια, μια, μια επανάσταση στην υγεία και το κλίμα. Για παράδειγμα, στις πόλεις της Ισπανίας, Βαλένθια, Μαδρίτη, γίνεται μία μετάβαση σε μία βιώσιμη μετακίνηση χωρίς καύσιμα, χωρίς ορυκτά καύσιμα. Για παράδειγμα, υπάρχει ένας, ε, ένας στόλ, θα έχουμε ένα στόλο ε, λεωφορείων καθαρά 100% ε, χωρίς, ε, ε, χωρίς ορυκτά καύσιμα του χρόνου. Αυτό είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει ολόκληρη η Ευρώπη. Είναι δυνατόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σβολικαν για ένα λεπτό από Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μεταφορέ στην Ευρώπη θα πρέπει να γίνουν πιο καθαρές και θα χρειαζόμαστε πιο φιλικέ προ το περιβάλλον όδους μεταφορά. Και νομίζω ότι είναι σωστό το γεγονό ότι με την οδηγία αυτή θέλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι οι δημόσιε προμήθειε θα δώσουν το καλό παράδειγμα. Κυρίως σε ό,τι αφορά τα λεωφορεία, γιατί οι δημόσιε μεταφορές αποτελούν 75% των, ε, οι δημόσιες μάλλον αγορές ε, το από πλευρά των κρατών αποτελούν 75% των ε, συνολικών και έτσι Στη Γερμανία έχουμε πολλά καλά παραδείγματα. Ε, το Βερολίνο μέχρι το 2030 θέλει να είναι χωρίς εκπομπές ε, μέχρι το 2030 και ήδη στην πατρίδα μου έχουμε ηλεκτρικά λεωφορεία, πιο πολύ από ό,τι σε όλη την υπόλοιπη Γερμανία. Όλα αυτά είναι εφικτά λοιπόν και γι' αυτό είναι σημαντικό και τα λεωφορεία με αέριο να αναγνωριστούν για ε, τα λεωφορεία στην καλεφορία που καλύπτουν μεγαλύτερε αποστάσει. Και νομίζω λοιπόν ότι κάνουμε ένα πολύ καλό και σημαντικό βήμα με την τρέχουσα νομοθεσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα η κυρία Σάλδεμούζα είναι η επόμενη ομιλήτρια για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αντιμετωπίζουμε πολλά κλιματικά προβλήματα και νομίζω ότι όλοι το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Όλοι όσοι παρακολουθούμε και τις εξελίξεις. Και χθες αυτό μας είπε και η Γκρέτα Τούνμπερκ. Έχουμε λοιπόν προβλήματα σε ό,τι αφορά και τις πολιτικές και σε ό,τι αφορά την ε, ρήπανση της ατμόσφαιρας που είναι πολύ φτωχή ποιότητα. Τα καθαρά οχήματα είναι τμήμα τη λύση, θεωρώ, και πραγματικά θα μπορούσαμε να έχουμε θέσει του στόχου σε πιο υψηλό επίπεδο, να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Παρ' όλα αυτά, κάτι κάνουμε τουλάχιστον τώρα θέτουμε δεσμευτικού στόχου για του Δήμου και τι κοινότητε σε ό,τι αφορά την πολιτική των δημοσίων συμβάσεων, τι αγορέ, τι δημόσιε των οχημάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν επιλύει το πρόβλημα τη ρήπανση τη ατμόσφαιρα, δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά τουλάχιστον είναι ένα σημαντικό βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Ελπίζω, ελπίζω το επόμενο κοινοβούλιο να δείξει πιο υψηλό επίπεδο φιλοδοξία από ότι και εμεί. Καλωσορίζουμε παρόλα αυτά το γεγονό ότι γίνεται μια βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Μπούλτς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Okay. Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Χαίρομαι που παρατηρώ πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί να στηρίζει ε, αυτή την πρόταση. Θέλω να ξαναευχαριστήσω τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές για τις επικοδομητικές διαπραγματεύσεις που μας επέτρεψαν να συμπληρώσουμε, να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία αυτή έγκαιρα πριν διακόψει το Κοινοβούλιο μαζί με, άλλα, μαζί με τα άλλα στοιχεία των πακέτων κινητικότητας 1, 2, 3, η αναθεωρημένη οδηγία θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο να μας βοηθήσει να πετύχουμε σημαντικές μειώσεις εκπομπών στον τομέα των μεταφορών που είναι απαραίτητες προκειμένου να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας με τη Συμφωνία COP29 του Παρισιού η υιοθέτησή της θα αποτελέσει έγκυρη, έγκαιρη συγγνώμη, συνεισφορά στην επιτεύξη αυτών των στόχων μέχρι το 2025. Πριν κλείσω, θα ήθελα όμως να κάνω ένα-δύο σχόλια στα όσα είπατε. Πρώτον, σε ό,τι αφορά το επίπεδο φιλοδοξίας μας. Πράγματι, αυτό το πακέτο, αυτή η πρόταση, είναι φιλόδοξη. Αλλά αυτό είναι που χρειαζόμαστε. Ακριβώς αυτό. Ταυτόχρονα είναι και ρεαλιστική. Και συνάδει με τις προβλέψεις για την αγορά. Να υπογραμμίσουμε ότι η πόλη γύρω τη σημαντικά δίκτυα δηλαδή πόλεων, ε, τοπικές, ε, η Local Governance for Sustainability, το Συμβούλιο Δήμων και Κοινοτήτων έχουν ε, εκφράσει και στο Κοινοβουλίο και στην Ρωμανική Προεδρία την πλήρη στήριξή του στην πρόταση της Κομισιόν. Οπότε ναι, ε, οι τοπικές κοινωνίες, οι τοπικές αρχές είναι έτοιμες. Οι... Τα οχήματα με μηδενικές εκπομπές αυτή τη στιγμή στηρίζονται σε... Ε, ε, έχουν ψηλή τιμή, αλλά αν το κόστος αυτό διαρρεθεί με το χρόνο ζωής τους, μειώνεται και θα μειωθεί ακόμα περισσότερο μέχρι να εφαρμοστεί η Οδηγεί αυτή, πολύ δε περισσότερο, που οι οικονομίε κλίμακο θα ρίξουν ακόμα περισσότερο το κόστο. Η οικονομική στήριξη είναι απαραίτητη, αλλά είμαστε διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουμε και υπάρχοντα ε, ε, χρηματοδοτικά όργανα όπως το Connecting Europe, Facility, ε, το EFSI κλπ. Να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει ένα κονδύλιο ακόμα και για τα ηλεκτρικά λεωφορεία, το οποίο ήδη χρησιμοποιείται από πολλές ε, ευρωπαϊκές πόλεις. Οπότε είναι σημαντική η σαφής στόχη για τις κρατικές προμήθειες και θα διευκολύνουν αυτή τη διαδικασία. Ένα σχόλιο τώρα σε ό,τι αφορά μάλλον κάποιες περισσότερες πληροφορίες για την αυτοκινητοβιομηχανία. Τον Ιούνιο του 2018 μια ομάδα μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών, Solaris, Skoda, Volkswagen, Ursus κλπ. έστειλαν μια ανοιχτή επιστολή στο Συμβούλιο και ζητούσαν περισσότερα φιλόδοξους στόχου από αυτούς που πρότεινε η Κομισιόν και επιβεβαίωναν ότι είναι έτοιμες να ανταποκριθούν. Οπότε ενθαρρυνόμαστε σε αυτή μας την ε, σε αυτήν την κατεύθυνση που κινούμαστε και από τις δύο πλευρές, και από τους αγοραστές και από τους πολιτές. Επίσης να επιβεβαιώσω αυτό που είπατε. Πολλές μεγάλες πόλεις ήδη έχουν ξεπεράσει τους στόχους σε ό,τι αφορά στις, ε, ε, στις ε, δεσμεύσεις τους. Ο στόχος της οδηγίας είναι να ενθαρρύνει και άλλες πόλεις να ακολουθήσουν αυτό το καλό παράδειγμα, αναγνωρίζοντας ότι πολλές μικρές και μεσαίες πόλεις ενδεχομένως δεν είναι ακόμα έτοιμες, δεν έχουν επαρκή τεχνογνωσία ή πόρους όπως το Άμστερνταμ ή το Παρίσι. Είμαστε όμως έτοιμοι να τις βοηθήσουμε για να διαπραγματευτούν από κοινού καλύτερες τιμές με την αυτοκινητοβιομηχανία. Οπότε αναμένω να υιοθετηθεί η έκθεση ε, του κύριου Ξιπ αύριο. Αυτό το θέμα, αυτό το κείμενο αποδεικνύει ότι αναγνωρίζουμε τη σαφή ανάγκη και ότι ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε σημαντικά ωφέλη για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Yes, Madam Ευχαριστούμε, κυρία Επίτροπε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα θετικά σας λόγια. Οπότε τώρα θα ακούσουμε τον εισηγητή μας, τον κύριο Ξύπα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο ηλεκτρισμός ως πηγή ενέργειας είναι πράγματι πολύ αποτελεσματική πηγή για τα αυτοκίνητα. Είναι βέβαια ακριβώς, ακριβή πηγή. Επίσης γνωρίζουμε ότι στηρίζοντας την ανάπτυξη του τομέα αυτού, δηλαδή των καθαρών οχημάτων, σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές και στην ε, παραγωγή, στην κατασκευή ε, οχημάτων. Πώς θα πείσουμε λοιπόν τον κόσμο εφόσον θα έχουμε πιο καθαρό αέρα, ατμόσφαιρα. Τα καθαρά οχήματα βοηθούν να έχουμε πιο καθαρή ατμόσφαιρα, άρα αυτό ακριβώς που θέλει ο κόσμος και ζητά. Και έχω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Υπάρχει ένας καθηγητής σε μια πολωνική πόλη που του αρέσει να τρέχει. Και μετά από πολλά χρόνια που έτρεχε είπε «Ξέρω ότι έχω κάνει κάτι στραβό, κάτι λάθος, γιατί τώρα έχω πρόβλημα με τα πνευμόνια μου». Αυτό δείχνει πόσο πολλοί είναι οι πολίτες που τελικά έχουν προβλήματα στην αναπνοή, πεθαίνουν πρόωρα εξαιτίας της ρήπανσης της ατμόσφαιρας. Όλο περισσότερες πόλεις βλέπουν τις αρχές τους να αποφασίζουν να περιορίζουν την πρόσβαση των οχημάτων στο κέντρο των πόλεων αυτών. Και τα μόνα οχήματα τα οποία επιτρέπονται είναι τα ηλεκτρικά. Και αντιλαμβάνομαι αυτό που είπε κάποιος νωρίτερα εδώ, ότι σίγουρα επιβάλλονται περιορισμοί από τις χώρες μέλη, από τις τοπικές αρχές, ε, σε μερικές περιπτώσεις, αλλά ε, δεδομένων των επαφών που έχω με την τοπική αυτοδιοίκηση σε περιφέρειες, πόλεις, δήμους κτλ. Πρώτα γίνονται διαβουλεύσεις και μετά λαμβάνονται αποφάσεις. Και βλέπω ότι ο κόσμος τελικά ε, θέλει να δεχτεί τον ευρύτερο ορισμό για οχήματα μηδενικών εκπομπών καθαρά οχήματα που κυκλοφορούν με μεθάνιο, με οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να προσαρμόσουμε επίσης τα που ήδη βρίσκονται στην αγορά. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία έχουμε αναπτύξει στις διαβουλεύσεις που έχουμε τους κοινωνικούς εταίρους και με τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, αλλά και άλλους ενδιαφερόμενους, κυρίως τις τοπικές αρχές, γιατί μας λένε τι περιμένουν να περιλαμβάνει η νομοθεσία αυτή προκειμένου να γίνει αποδεκτή. Εννοείται ότι πρόκειται για ένα συμβιβασμό μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων του Κοινοβουλίου, ε, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε θέλω να εκφράσω εδώ τις ευχαριστίες μου σε όσους συμμετείχαν στην εκπόνηση αυτού του κειμένου. Αυτό που πρέπει επίσης να γνωρίζετε είναι ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια μετά το 2020 θα στηρίξουν τους στόχους της οδηγίας. Και είναι και αυτό ένα κίνητρο για εκείνους που θέλουν να εμπλακούν στην υλοποίηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για τη συνεργασία σας, όλους σας, για τη συνεργασία σας όχι μόνο στην οδηγία αυτή ε, και σας, γιατί όλοι μαζί συνεργαζόμαστε για να πετύχουμε κάτι. Δεν συμφωνούμε πάντα όλοι σε όλα, αλλά πιστεύουμε όλοι ότι κάνουμε κάτι καλό για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Η ψηφοφορία για το θέμα αυτό θα λάβει χώρα αύριο. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μπούλτς για την παρουσία της εδώ. Καλό σας βράδυ. Και καλωσορίζω εδώ την κυρία Γιούροβα, την Επίτροπο Γιούροβα και θα συζητήσουμε τώρα μαζί της την έκθεση του κυρίου Ταντέου Σβιεφκά πρόκειται για την χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου. Η έκθεση του κ. Ζιέφκα. Έχετε το λόγο κ. Ζιέφκα. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να απευθυνθώ σε εσά, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, βλέπουμε ότι η θητεία ολοκληρώνεται, αλλά υπάρχουν ακόμα αρκετά σημαντικά θέματα τα οποία και πρέπει να εγκρίνουμε. Η ευρωπαϊκή αγορά, οι επιχειρήσει στην Ευρώπη περιμένουν και θα ήθελα ευθύ εξ αρχή ε, να ευχαριστήσω την κυρία Επίτροπο, την κυρία Γιούροβα, ε, Επίσης, να ευχαριστήσω την ομάδα της γιατί ε, έκαναν ε, πάρα πολύ καλή δουλειά, ε, κατέθεσαν μια θαυμάσια πρόταση και έτσι περιόρισαν και το χρονικό διάστημα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τέστη λοιπόν δυνατόν να διεξάγουμε τις διαπραγματεύσεις στον τριμερή διάλογο με απόλυτη ηρεμία και ησυχία. Ευχαριστώ τους και τις εισηγήτριες, τους συναδέλφους μάλλον, που ήταν σκιώδη εισηγητές. Περί πρόκειται, πρόκειται για το εταιρικό δίκαιο που είναι πολύ σημαντικό για την κοινή αγορά. Και πρόκειται κατ' ουσίαν και για ένα πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί την κοινωνία, την ψηφιοποίηση. Η νέα οδηγία δίνει νέες δυνατότητες για την καταχώρηση των επιχειρήσεων, όπου ε, μπορεί κανείς να εκμεταλλευτεί τις ε, ψηφιακές ε, τεχνολογίες, συγκεκριμένα το διαδίκτυο. Είναι βέβαια λίγο περίεργο το ότι μόνο στο τέλος της θητείας συζητάμε για την ψηφιοποίηση σε σχέση με τα δικά μας τα θέματα για την ε, κοινωνία της πληροφορίας. Μιλάμε αρκετό καιρό, αλλά τώρα αυτό που ενδιαφέρει είναι το τι προσδοκούν οι εταιρείε από εμάς. Κυρίες και κύριοι, ένα πράγμα είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ο στόχος που έχουμε είναι η βελτίωση, η διευκόλυνση της ζωής των εταιριών σε αυτό το θέμα της ε, καταχώρησής τους. Πρόκειται για έγγραφα, παραστατικά, το πώς ε, διαβιβάζονται, ε, το πώς γίνεται ο συντονισμός ανάμεσα στα διάφορα κρατημέλη. Βέβαια υπάρχουν ήδη αυτές οι δυνατότητες, αλλά η όλη διαδικασία ήταν χρονοβόρα και δαπανηρή. Και η υπάρχει και μια ανασφάλεια σχετικά με το πώς γίνεται η καταχώρηση σε ένα άλλο κράτος μέλος. Έτσι λοιπόν προέκυψε το εξής. Οι δυνατότητες στην αγορά εξαφανίστηκαν ή εξαφανίζονται πριν καν δραστηριοποιηθεί μια εταιρεία. ή δεν υφίστατο καθόλου ή ήταν αναγκασμένη να παραιτηθεί από συμβάσει γιατί ο χρόνο για καταχώρηση ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Τώρα λοιπόν με αυτή την πρόταση περιορίζουμε το χρόνο καταχώρησης, η ψηφιακή καταχώρηση πρέπει να, μπορεί να γίνεται από 5 μέχρι το πολύ 10 ημέρες. Βεβαίως ε, πρέπει να εκπληρώνονται όλες οι υποχρεώσεις, ε, ε, πρέπει να κατατίθενται όλα τα απαραίτητα έγγραφα και βεβαίως στην οδηγία εκφράσαμε κάποιες ε, επιφυλάξεις για την αντιμετώπιση του ενδεχομένου απάτης. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με τα θέματα που συζητάμε. Κυρίες και κύριοι, πολύ συγκεκριμένα, για ποιες επιχειρήσεις πρόκειται, έχω στοιχεία που δείχνουν ότι έχουμε περίπου 24 εκατομμύρια εταιρείες στην Ευρώπη και περίπου το 80% εξ αυτών είναι κεφαλαιακές εταιρείες και οι περισσότερες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι εκείνες που προσφέρουν και τις περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Εάν λοιπόν διευκολύνουμε τη δική του τη λειτουργία, ε, ξεκονομώντας χρόνο, χρήμα, προσωπικό, αυτό θα είναι πολύ σημαντικό και ακριβώς αυτό θέλουμε να επιτύχουμε με την έκθεσή μας. Οι διατάξεις αφορούν, όπως σας είπα, κεφαλαϊκές εταιρείε. και τώρα απευθύνομαι στην Επίτροπο, την κυρία Γιούροβα και θέλω να της πω ότι κατά τον έλεγχο που θα γίνει μετά από έξι περίπου χρόνια, κατά την αναθεώρηση, όλο αυτό το θέμα, η ψηφιακή καταχώρηση θα πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις εταιρείε. Κυρίε και κύριοι, υπάρχει ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό για εμένα το ότι είναι απαραίτητο να συνεργάζονται τα κράτη-μέλη σε ορισμένα θέματα, περί ποιων θεμάτων ομιλώ ή σε ποια αναφέρομαι. Αναφέρομαι, παραδείγματο χάρη, στα θέματα της ε, διαχείρισης, ε, στις ηγετικέ θέσεις, ε, κατά πόσον κάποιος μπορεί να αναλαμβάνει μία ηγετική θέση σε μία εταιρεία. Είναι λίγο περίπλοκο αυτό και για το λόγο αυτό παρατείνουμε και τον χρόνο εφαρμογής της οδηγίας. Βεβαίως μπορεί κανείς να σχιστεί ότι αυτό περιπλέκει περαιτέρω την κατάσταση, αλλά σε τελική ανάλυση νομίζω ότι απορρέει όφελος ε, για όλα τα κράτη-μέλη. Ε, αν υπάρχει σωστή εφαρμογή, σύντομα προκύπτει και όφελος. Και νομίζω ότι αυτό θα το εσαρτούν οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν καλώ όλους σας αύριο να εγκρίνει το θέμα κατά την πρώτη ανάγνωση. Ευχαριστώ η κυρία Γιούροβα. Αύριο θα μετακινηθούμε, θα κινηθούμε ένα βήμα πιο κοντά στο να φέρουμε την νέα αγορά στις ε, εταιρείε. Και όπως είπε και ο συγγετής, ε, είναι η τελευταία μας ευκαιρία θα βοηθηθούν οι επιχειρηματίες ε, να δικούν πιο εύκολα και πιο φτηνά τις επιχειρήσεις. Θα έχουμε επιγραμμικές διαδικασίες τώρα σε όλα τα κράτη-μέλη. Οι εταιρείε θα μπορούν να χρησιμοποιούν πλήρως ε, τα ψηφιακά εργαλεία και στις διαδικασίες όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και διασυνοριακά. Οι εταιρείε θα σώζουν χρόνο και χρήμα όταν θα ιδρύουν μία νέα επιχείρηση υποκατάστημα και θα έχουν διαθέσιμε πληροφορίε στα επιχειρηματικά μητρώα. Και όλα αυτά με τα υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή, τον κύριο Τσβιέφκα, και τις Προεδρίες του Συμβουλίου για την ταχύ εργασία τους επί της πρότασης και για την εξαιρετική συνεργασία. Η Κομισιόν είναι ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα. Ιδίω η πολιτική συμφωνία για την οδηγία για τα ψηφιακά εργαλεία και τι διαδικασίε αποσαφηνίζει περαιτέρω ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να διατηρήσουν τα εθνικά του εφιστάμενα συστήματα, τι απαιτήσει και τι διαδικασίε, ενώ θα καταστήσουν δυνατέ τι επιγραμματικέ διαδικασίε για τη σύσταση των εταιριών, την καταγραφή υποκαταστημάτων και την κατάθεση εγγράφων. Ως σημαντική ασφαλιστική δικλίδα κατά της απάτης, η οδηγία θα διευκρινίσει σε ποιες ε, ε, εξαιρετικές περιπτώσεις τα κράτη-μέλη μπορούν να απαιτούν φυσική παρουσία στις διαδικασίες. Επίσης, χαίρομαι που οι συνομοθέτες συμφωνήσαν για τους κανόνες που αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών για τους αποκλεισμένους διευθυντές. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση ενός πιο διαφανούς επιχειρηματικού περιβάλλον και την καταπολέμηση της απάτης. Επίσης, περισσότερες πληροφορίες από τα επιχειρηματικά μητρώα θα είναι δωρεάν διαθέσιμες στα ενδιαφερόμενα μέρη κυρίως για το ποιος νόμιμα μπορεί να εκπροσωπήσει μια εταιρεία. Αυτό θα συνεισφέρει στο να υπάρχει περισσότερη εμπιστοσύνη στις επιχειρηματικές συναλλαγές. Η Κομισιόν υποστηρίζει πλήρως το συμβιβασμό που βρήκαν οι συνομοθέτες και ανυπομονή για την ευριανή ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος του ΕΛΚ, ο κύριος Ράντεφ, για μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για τη συμφωνία και την τελική εκδοχή του κειμένου. Η οδηγία θα ωφελήσει καταρχήν τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Ε, η έλλειψη κανόνων εγγραφής online και οι αποκλήσεις μεταξύ των κρατών μελών ε, προκαλούσαν ε, γραφειοκρατία και το κόστος για όσους ήθελαν να ιδρύσουν μια εταιρεία ή να αναβαθμίσουν τη δραστηριότητά τους μέσω μιας, ενός υποκαταστήματος ή μιας θεγατρικής αλλά μέλη. Τώρα, θα έχουμε πιο εύκολους ε, κανόνες για την εγγραφή των εταιριών περιορισμένης ευθύνης. Τα έγγραφα θα μπορούν ε, να σταλούν ε, επιγραμμικά στο Μητρό. Η επιγραμμική εγγραφή είναι πιο φθηνή και η Βουλγαρία έχει εισαγάγει αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει πιο γρήγορη διεκπαιρέωση των εγγράφων και φυσικά δεν σημαίνει αυτό ότι θα έχουμε υψηλότερο κόστος ε, με την ε, επιγραμμική εγγραφή. Είναι πολύ σημαντική και η αρχή άπαξ μόνον. Η εταιρεία θα πρέπει μόνο μία φορά να παρέχει ορισμένες πληροφορίες. Η επιγραμμική εγγραφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ωφελήσει πάρα πολύ τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι ψηφιακές λύσεις, το εταιρικό δίκαιο προσφέρουν υψηλά ποιότητα προστασίας, ελέγχους ταυτότητας ε, και πιθανές ε, ε, συνεντεύξεις με παρουσία είναι κάποια από τα κύρια στοιχεία της πρότασης. Οι πληροφορίες για τις εταιρείες θα είναι δυνατόν, θα είναι προσβάσιμες και αυτό θα είναι πολύ μεγάλο όφελος για τις εταιρείες. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρέγνερ έχει το λόγο. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε Ισηγητά, με την ψηφιοποίηση των εταιριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο μέλλον οι εταιρείε θα μπορούν να συστήνονται επιγραμμικά, να κατατίθενται τα έγγραφα επιγραμμικά και όλες οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται επίσης επιγραμμικά. Οι προϋποθέσεις βεβαίως παραμένουν σε εθνική αρμοδιότητα. Η δική μου η πολιτική ομάδα δεν ήταν εκ των προτέρων σύμφωνη, γιατί για τους σοσιαλδημοκράτες είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ισχύουν αυστηρές προδιαγραφές κατά των απατών, ε, όταν δηλαδή τα κράτη δίνουν τη δυνατότητα σε εταιρείε να συστήνονται με ένα απλό πάτημα του ποντικού. Εμείς δεν θέλουμε να υπάρχουν εικονικές εταιρείε, ούτε να προάγουμε επιχειρηματικά μοντέλα που ε, ορίζονται ως το Delaware της Ευρώπης. Γι' αυτό λοιπόν ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο εισηγητή, την κυρία Επίτροπο, συγχαρητήρια στην διαπραγματευτική ομάδα, στην Σκιώδη εισηγήτρια, ε, το αποτέλεσμα προβλέπει το εξή. Η δεσμευτική, ο δεσμευτικό έλεγχο τη ταυτότητα των ανθρώπων που θέλουν να συστήσουν την εταιρεία ε, τα κράτη-μέλη παρά την πλήρη ψηφιοποίηση για λόγους δημοσίου δικαίου μπορούν να καλέσουν αυτά τα άτομα να παρουσιαστούν στην αρμόδια υπηρεσία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό έτσι ώστε η επιγραμμική καταχώρηση να μην γίνει ένα εργαλείο για εικονικές εταιρείε. Νέε λοιπόν προϋποθέσεις, καλύτερη πληροφόρηση, αυτά θα πρέπει να φαίνονται από τα μελλοντικά λογιστικά στοιχεία για να μπορεί να λειτουργεί και το σύστημα BRIS. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι στο μέλλον σε όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εισαχθούν κανόνες έτσι ώστε να αποκλείονται κάποια στελέχη από τις εταιρείε, οι απαταιώνες θα πρέπει να μπορούν να εξαπατούν ε, άλλα κράτη-μέλη. Οι επιχειρήσεις ε, θα πρέπει να μπορούν να εκμεταλλεύονται την ψηφιοποίηση, αλλά η Ευρώπη δεν θα μπορεί να γίνει ένα σούπερ μάρκετ ε, ψηφιοποίησης με τις αυστηρές προδιαγραφές και με τον έλεγχο της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου. Τα κράτη-μέλη θα μεριμνούν έτσι ώστε να μην προκύπτει κατάχρηση του εταιρικού δικαίου. Συγχαρητήρια λοιπόν για το σπριντάρισμα, θα το χαρακτηρίσω αν μου επιτρέπετε, το οποίο κατορθώσαμε έστω και στο τέλος της θητείας αυτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε. Επόμενος πακέτ εκ μέρου του ECR. Έχετε το λόγο. 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Στην Φλάνδρα οι μικρομεσές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν και τη σποδηλική στήλη της οικονομίας. Ε, ζούνε χιλιάδες και χιλιάδες οικογένειες από αυτές. Τώρα μιλάμε για την ψηφοποίησή τους. Και μιλάμε και για το δίκαιο που όντως πρέπει να συνοδεύει αυτή την ε, ψηφιοποίηση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός και για να συμβεί αυτό πρέπει οι χώρες μέλη να φροντίσουν η ψηφιοποίηση αυτή να γίνει όσο γίνεται πιο απλά. Οι δυνατότητες μιας επιχειρίας να οργανωθεί ψηφιακά δεν πρέπει να επιτρέπει κανένα περιθώριο απάτης. δεν ε, θα πρέπει να υπάρχουν παραθυράκια ώστε να μπορεί να γίνεται νομιμοποίηση, για παράδειγμα, παράνομου χρήματος. Πρέπει να βρεθούν τα μέσα εκείνα τα οποία θα εγγυηθούν για την ασφάλεια, μέσα για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση ή οτιδήποτε άλλο για την καταχώρηση στο Μητρό. Όντω, για τι επιχειρήσει τα πράγματα πρέπει να γίνονται πιο εύκολα, πιο απλά. Πρώτα απ' όλα γιατί έτσι εξοικονομούν χρήματα, αλλά και γιατί θα μπορέσουν να δημιουργηθούν και περισσότερε επιχειρήσει. Και αυτό σίγουρα θα είναι θετικό, εφόσον θα γίνεται ηλεκτρονικά η καταχώρησή του. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Σφιέσκα για να κλείσει τη συζήτηση, προηγουμένως η Επίτροπος έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρεμβάσεις σας όλους και πράγματι σας ενθαρρύνω να υπερψηφίσετε το κείμενο αυτό, αυτή την πρόταση. Με την νομοθετική αυτή πρόταση, όντως, καλούμε τις μικρομεσαίες και γενικά τις επιχειρήσεις στον 21ο αιώνα είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Κάνουμε κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Επίσης, μπορούμε τώρα να επικεντρώσουμε και τις προσπάθειές μας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η υλοποίηση ε, θα γίνει εφικτή και στην πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή για τις τελευταίες του σκέψεις από αυτού και συγχαρητήρια και για το έργο σας, έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω κι εγώ να ευχαριστήσω την Επίτροπο και όλους τους συναδέρφους για τη συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι ολοκληρώνεται έτσι μια μεγάλη διαδικασία συνεργασίας κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας. Για μας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Συνομοθέτης, είναι προφανές ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις αποτελούνται από ανθρώπους με κυριότητα, οι οποίοι δεν θα προβούν σε απάτες. Προτείνουμε λοιπόν καλές λύσεις για να διευκολύνουμε την καθημερινότητά τους. Η καθημερινότητα είναι ψηφιακή έτσι καλλιώ σήμερα. Απάτες πάντα συνέβαιναν και πάντα θα συμβαίνουν. Και στην κλασική καταχώρηση δεν βλέπω γιατί τώρα να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες για απάτες. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στις εργασίες μας και συνεισέφεραν επενδύοντας χρόνο και έργο για να ετοιμαστεί αυτή η νομοθετική πρόταση. Και προς το Συμβούλιο θέλω να πω ότι δεν πρέπει να αργήσουμε να εφαρμόσουμε την οδηγία αυτή. Οι πολίτες μας περιμένουν ανυπόμονα αυτό το νομικό μέσο που είναι τόσο σύγχρονο και ελπίζω αυτό να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε εδώ τη συζήτηση. Αύριο θα έχουμε την ψηφοφορία για την έκθεση αυτή. Στη συνέχεια, αγαπητοί συνάδελφοι, στην Μυρσή διάταξη έχουμε την έκθεση τη κυρία Εύελιν Ρέγκνερ, Διασυνοριακέ μετατροπέ Συγχωνεύσει και διασπάσει. Καταρχήν, θα ακούσουμε την εισηγήτρια για τέσσερα λεπτά. Αξιότιμη κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Αυτό το οποίο καταφέραμε εδώ είναι ένα ορόσημο. Η οδηγία είναι περίπλοκη, είναι πολύ διευρυμένη, έχει σχέση και μπορεί να συγκριθεί με την οδηγία περί προστασίας δεδομένων, παραδείγματο χάρη, σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορέσαμε να συνδυάσουμε την εντολή των δύο θεσμών και να επεξεργαστούμε ένα κοινό κείμενο. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους, την Επιτροπή, ε, την Επίτροπο, τους και ηγητές, αλλά και το Συμβούλιο. Έχουμε λοιπόν ένα νέο ε, νόμο ο οποίος ε, προβλέπει και ρυθμίζει την κινητικότητα των επιχειρήσεων και εισάγει μια ενιαία διαδικασία για τις ε, συγχωνεύσεις και τις διασπάσεις των εταιριών. Ναι, πράγματι όλες οι εταιρείε έχουν το δικαίωμα να μετεγκαθίστανται σε μια άλλη χώρα. Εγώ Προέρχομαι από τα συνδικάτα και θεωρώ ότι τα οι εταιρείε θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να μετακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο που αυτό το δικαίωμα ποτέ δεν απέτυχε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Γι' αυτό λοιπόν ε, ισχύει η νομολογία, αλλά η νομολογία ήταν πέρα από τους νόμους και αυτό έδωσε τη δυνατότητα στο να δημιουργηθούν εικονικές εταιρείε. Γι' αυτό εμένα αυτό που ενδιαφέρει είναι να υπάρχει μια ισορροπία. Οι εταιρείε μπορούν να ασκούν ε, το δικαίωμά τους, αλλά όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, κυρίως οι εργαζόμενοι, θα πρέπει να είναι σωστά προστατευόμενοι. Μπορέσαμε να βρούμε έναν καλό κοινό παρονομαστή. Οι βασικέ προποθέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εμφανίζονται σε αυτή τη νέα οδηγία. Καλύτερη προστασία των εργαζομένων όταν τα κράτη-μέλη μετακινούνται σε άλλο κράτο μέλο. Και επίση ε, και μια δεσμευτική ρήτρα κατά των καταχρήσεων ε, για να μπορούμε ακριβώ να αποφύγουμε αυτέ τι εικονικέ εταιρείε. Ε, το θέμα του προσωπικού με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να εισακούνται, να ενημερώνονται όταν πρόκειται για την ύπαρξή τους και για, ε, και για την εργασία τους. Η σωστή ενημέρωση των εργαζομένων επιτρέπει στο μέλλον να είναι δικαίωμα η ενημέρωση των εργαζομένων για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Να υπάρχει δεσμευτική, υποχρεωτική, να υπάρχουν υποχρεωτικά διαβουλεύσεις και επιπλέον εισάγονται και νέα ε, δικαιώματα για τους εργαζόμενους ε, όταν μια χώρα μετεγκαθίσταται. Ε, οι εργαζόμενοι στο μέλλον θα έχουν μια εκτενή έκθεση στα χέρια τους για το μέλλον των θέσεων απασχόλησής τους, θα ερωτώνται για τη μετεγκατάσταση, θα μπορούν έγκαιρα να τοποθετούνται και για πρώτη φορά αποκτούν το δικαίωμα να ζητούν αιτιολογημένη άποψη από την διοίκηση. Επίσης, καθίσατε σαφές ε, ότι οι εθνικοί κανόνες οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους ε, τις, ε, τους ενωσιακούς κανόνες και επίσης το ότι τα εργοστασιακά συμβούλια θα πρέπει να έχουν επαρκείς πόρους για να μπορούν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Το θέμα του συναποφασίζει, βελτιώνεται με την πρόταση της Επιτροπής και εδώ προβλέπεται προστασία τεσσάρων ετών και αυτό ισχύει για ε, ορισμένα, για όλα τα κράτη-μέλη κάτω βέβαια από ορισμένε προποθέσει. Ο δεύτερο τομέα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ απορρέει από την εργασία που έκανα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα ε, φορολογικά σκάνδαλα, τα LuxLeaks, ε, τα Panama Papers και πολλά συναφή όσον αφορά την απόσπωση των εργαζομένων, κυρίω στον τομέα των μεταφορών. Εκεί υπάρχουν πολύ συχνά καταχρήσει μέσω των εικονικών εταιριών. Το εταιρικό δίκαιο συστηματικά είναι αντικείμενο καταχρήσεων για να βρουν ενδιαφερόμενοι τις καλύτερες συνθήκες, ε, συνήθως εις βάρος στην πλάτη των εργαζομένων. Γι' αυτό λοιπόν είμαι πολύ υπερήφανη για μια δεσμευτική ρήτρα κατά των καταχρήσεων που προβλέπεται πλέον η αρμόδια υπηρεσία στην οποία το δικαστήριο πρέπει να απευθυνθεί. Εάν η αρμόδια υπηρεσία υποπτεύεται ότι υπάρχει κατάχρηση, πρέπει να εξετάσει στις τρεις υποχρεωτικές διαδικασίες ε, κατά πόσον πράγματι τηρήθηκαν τα εθνικά και τα ε, ενωσιακά δικαιώματα, μήπως έγιναν κάποιες προσπάθειες παράκαμψή τους ή μήπως υπάρχουν άλλοι εγκληματικοί στόχοι. Εάν διαπιστωθεί ότι ισχύει κάτι από όλα αυτά, τότε δεν θα δίδεται η άδεια σε μία εταιρεία. Εάν λοιπόν μία εταιρεία τελήσει, να παρακάμψει δικαιώματα ή να συστήσει παράνομα εικονικές εταιρείε, τότε η μετεγκατάσταση απαγορεύεται. Αυτή λοιπόν η ρήτρα που ισχύει και για συγχωνεύσεις και για διαιρέσεις εταιριών, αυτή η συγκεκριμένη ε, οδηγία παίρνει σάρκα και οστά. Εάν μετά την αναδιάρθρωση προκύψουν ύποπτες εξελίξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να επιβάλλουν πρόστιμα. Με την κινητικότητα των εταιριών δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν πλέον καταχρήσεις και εικονικές εταιρείε. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα εκτεταμένο πακέτο, μία δέσμη μέτρων που μου επιτρέπει να ευχαριστήσω όλους τους και οδησηγητές, τον κύριο Ντεγκράντε και τον Πασκάλ Ντιγόν, οι οποίοι όλοι προσπάθησαν αυτή την ε, εκτεταμένη δέσμη μέτρων επιτέλους να την ε, καταστήσουν σε κάτι το απόλυτα συγκεκριμένο. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιούροβα έχει το λόγο εξ ονόματο της Επιτροπής Αξιότιμα Μέλη του Κοινοβουλίου. Θα ξεκινήσω την ομιλία μου με συγκίνηση, γιατί είναι η τελευταία ολομέλεια για μένα στη θητή αυτή. Συμμετείχα σε τόσες ε, πολλές ε, την τελευταία πενταετία και πρέπει να πω ότι εργαστήκαμε για πάρα πολλά θέματα και με την κυρία Ρέγνερ και με τον κύριο Ντεγκράντες και πάντοτε αισθανόμουν ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη η συνέργεια πολιτικής βούλησης, ε, λογικής ε, και κατανόησης. Και νομίζω ότι αυτό αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα, αυτό το πακέτο εταιρικού δικαίου, ε, που είναι πολύ πολύπλοκο, αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα. Και Πολλοί δεν πίστευαν ότι θα τα καταφέρναμε να το ολοκληρώσουμε. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο τέλος μιας πολύ δύσκολης αλλά επιτυχούς διαδικασίας. Η Ευρωπαϊκή Αγορά προσφέρει πολλές ευκαιρίες στις εταιρείε ε, να αναπτυχθούν. Όμω, πολύ συχνά οι εταιρείε ε, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα ωφέλη στην πράξη. Η πρόταση τη Κομισιόν απάντησε ε, σε αίτημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα συνδικάτα και τι οργανώσει των επιχειρήσεων για νέου κανόνε στον τομέα αυτό. Και θέλω να ευχαριστήσω την συγγήτρια, την κυρία Ρέγνερ ε, και τι αντίστοιχε προεδρίε του Συμβουλίου για την επικοδημητική του προσέγγιση και την αποτελεσματική του δουλειά σε αυτή την ιδιαίτερα πολύπλοκη και σημαντική σημαντική πρόταση. Χαίρομαι πολύ που το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρήκαν ένα ρεαλιστικό και καλό συμβιβασμό που θα βελτιώσει σημαντικά την κατάσταση και για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους υπαλλήλους. Η οδηγία θα βοηθήσει τις εταιρείε ε, να μετακατασταθούν και να οργανωθούν στην ενιαία αγορά, ενώ θα παρέχει τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλίδες για τους ε, ενδιαφερομένους και τους υπαλλήλους η Κομισιόν. Καλωσορίζει τον ε, υποχρεωτικό χαρακτήρα των μέτρων κατά της κατάχρησης. Ήταν ένα σημαντικό θέμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για πολλά από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Κομισιόν καλωσορίζει επίσης τις διατάξεις για τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπου περιλαμβάνονται πολλά από τα θέματα που τέθηκαν στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το κατόφλι των τεσσάρων πέπτων για την έναρξη των διαπραγματεύσεων ε, και Στι ε, τρει διασυνοριακές πράξεις, ο υποχρεωτικό χαρακτήρας αυτών των διαπραγματεύσεων και οι διατάξει προστασία τη διαπραγματευόμενης λύση. αν ε, ε, υπάρχουν και μετέπειτα πράξει, παρέχουν ένα πλήρε πακέτο ασφαλιστικών δικλείδων. Επιπρόσθετα, το νέο άρθρο για την ενημέρωση και την παροχή συμβουλών και τη διαβούλευση τονίζει και τα δικαιώματα των υπαλλήλων να έχουν λόγο σε μια διασυνοριακή διαδικασία. Και αυτό ήταν ουσιαστικό για το Κοινοβούλιο. Ε, θυμόμαστε τι αποκλίνουσε θέσει που υπήρχαν όταν ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσει. Και η Κομισιόν θα ήθελε να συγχαρεί του συνομοθέτε για τι λύσει ε, που βρέθηκαν ε, για ε, τον συμβιβασμό που αποτελεί ένα καλό βήμα προς τα μπρος σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση. Παρέχει εύρωστους και δίκαιους κανόνες για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ε, που συμμετέχουν σε συνοριακές διαδικασίες, ενώ δεν είναι πολύ βαριά η διαδικασία στην πράξη. Επομένως, η Κομισιόν μπορεί να υποστηρίξει πλήρως το συμβιβασμό και ανυπομονή για την αυριανή ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της ΕΚΟΝ, ο κύριος Λούντβικσον, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ήμουν συντάκτης γνωμοδότησης από πλευράς της Οικονομικής Επιτροπής και ετοίμασα την γνωμοδότησή μου που λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ασφαλείς κανόνες οι οποίοι να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να μετακινούνται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις επιχειρήσεις που εργάζονται σοβαρά. Συγχρόνως όμως χρειαζόμαστε και κανόνες που θα μας επιτρέψουν να καταπολεμήσουμε το dumping ε, στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα. Πρέπει να αποφύγουμε απλώς και μόνο ε, ο στόχος της μετακόμισης να είναι να αποφεύγονται οι κοινωνικοί κανόνες, δηλαδή να μην σεβόμαστε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστώ την εισηγήτρια την κυρία Ρέγνερ και όλους τους κοιόδης εισηγητές και όσους γνωμοδότησαν για την καλή συνεργασία που είχαμε μεταξύ μας και με το Συμβούλιο. Οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν τώρα περισσότερες δυνατότητες για ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσα στην εσωτερική αγορά. Συγχρόνως οι νέοι κανόνες προσφέρουν και μία ενισχυμένη ασφάλεια τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους μετόχους των επιχειρήσεων. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό αύριο να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε μεταξύ μας και είναι επίσης σημαντικό να έχουμε ασφαλείς κανόνες όταν πρόκειται για τα δικαιώματα των επιχειρήσεων μέσα στην εσωτερική αγορά. Συγχρόνως όμως να αποφύγουμε κάθε κατάχρηση, κάθε απάτη είναι πολύ σημαντικό γιατί αλλιώς θα υπονομευθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην εσωτερική αγορά. Μέσα από το κείμενο αυτό είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε περισσότερη δικαιοσύνη στην ενία αγορά. Είναι μια δικαιοσύνη η οποία θα επιτευχθεί εάν πάψουν να υπάρχουν εικονικές επιχειρήσεις. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ε, ξεκινάμε με τις πολιτικές ομάδες. Ο κύριος Δεγκράντες Πασκουάλ πρώτα απ' όλα εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Γιούροβα. Κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ το Συμβούλιο για το έργο του. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια και φίλη μου, αν και αντίπαλος πολλές φορές, την κυρία Ρέγνερ. Εμείς στο ΕΛΚ στηρίξαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή την οδηγία, γιατί ο κύριο στόχο είναι να διευκολύνεται η ζωή των επιχειρήσεων, των μικρομισών κυρίω, και να μπορούν ελεύθερα να μετακινούνται μέσα στην Ευρώπη. Θέλουμε ένα νομικό πλαίσιο μέσα σε ένα κόσμο όλο και πιο περίπλοκο, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για τους εργαζόμενους, τους μετόχους κλπ. Και γι' αυτό οι νέες εναρμονημένες διαδικασίες περιλαμβάνουν και τις ρήτρες ασφάλειας για να ε, σεβόμαστε και να προστατεύουμε τα δικαιώματα όλων αυτών. Κυρίε και κύριοι, έπρεπε να δώσουμε μια απάντηση μετά από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την ελευθερία εγκατάσταση. Βάσει του άρθρου 49 τη συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί πάντα υποστηρίζαμε ότι επιχειρήσει οι οποίε εγκαθίστανται σε μια χώρα μέρο έχουν το δικαίωμα και την ελευθερία να μπορούν να μεταφέρουν την έδρα του σε άλλη χωρί να χάνουν την νομική του προσωπικότητα. Αυτό το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί Μερικέ φορέ ακόμα και χωρί οικονομική δραστηριότητα στη νέα χώρα. Θεωρούμε όμω σημαντικό, όπω και η και το Συμβούλιο, να βάλουμε και μία ρήτρα κατά των καταχρήσεων. Όταν γίνονται τέτοιε διασυνοριακέ μετακίνησει, πρέπει να αποφεύγουμε απάτε και κατεχρήσει του συστήματο. Γι' αυτό λοιπόν εγώ προσωπικά, όπως ξέρει και η συγγήτρια, υπογράμμισα πάρα πολύ ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δικαιολογούνται. Δηλαδή, αν έχουν πάρει ε, κρατικές επιδοτήσεις, αν έχουν οικονομική ενίσχυση. Δεν μπορούν να φύγουν από τη χώρα, να υποφελούνται δηλαδή από το σύστημα και να αφήνουν ξεκρέμαστους και τους εργαζόμενους. Αυτό θέλουμε και στην Ισπανία. Εμείς επίσης θέλουμε ex post έλεγχο της μετακίνησης για να επαληθεύουμε ότι δεν υπάρχει καμία απάτη και να επικυρώνεται η δραστηριότητα αυτή μόνο εφόσον υπάρχει κατάλληλη εγγύηση για όλους. Το αποτέλεσμα πιστεύω ότι είναι θετικό. Υπάρχει ελευθερία μετακίνηση που ήταν πάντα η προτεραιότητά μα, γιατί πιστεύουμε σε μια ενωμένη Ευρώπη χωρί σύνορα. Αυτό είναι η προτεραιότητά μα και αυτή είναι και η ευθύνη μα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τεγκράντε Πασκουάλ. Τώρα, ε, για τους σοσιαλιστές, ο Μικαέλα Ντέτζεν. Δύο λεπτά. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε Επίτροπε, με την αυρινή ψηφοφορία ε, δίνουμε τέλος σε μια παράδεκτη κατάσταση όπου οι εταιρείε θα μπορούσαν να μετακινηθούν σε μια